Ο Πρόεδρος. Ε, Znawiam posiedzenie. Ε, witam wśród nas pana. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζωζεύ Μανουέλ Μπαρόζο. Πριν αρχίσουμε όμως την ώρα των ερωτήσεων θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια προς τα πρακτικά. Εάν όχι, εγκρίνονται. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Καλωσορίζω για μία ακόμα φορά τον κύριο Μπαρόζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.